Dear colleagues, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, We will start... θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. After suspension. Μετά τη διακοπή. Please take your seats. Καθίστε σας παρακαλώ. Uh, Έχω ανακοίνωση να σας κάνω. Μάμο Σας παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ. Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα. Υπάρχει μια γραπτή δήλωση υπεριθμών 26 κάθετος 2011, την οποία έχει υποβάλει μια σειρά βουλευτών, Σάρπο, Γέγκλε, Ιρουέρα, ε, Ρωμέβα, Ιρουέδα και άλλοι για τη διαχείριση των πληθυσμών σκύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου έχει υπογράψει και σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού θα διαβιβαστεί αρμοδίως και θα δημοσιευτεί στα κείμενα που θα εγκριθούν στη σημερινή συνεδρίαση θα επισυναυτούν και στα πρακτικά τα ονόματα των υπογραφών Και θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Σάρπου να πάρει το λόγο, που είναι εκ των συντακτών της γραπτής δήλωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους Βαλεάνου, Γέγλε, Βοητσεκόφσκι και Ρωμέβα Ιρουέντα για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν και τους υπολείπους συναδέλφους για τις υπογραφές τους χάρη σε αυτού το θέμα των αδέσποτων σκύλων μπορεί να βρει μια λύση. Ε, Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε και παίρνουμε στις ψηφοφορίες. Το πρώτο θέμα είναι